Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε και εγώ θα μιλήσω στα ισπανικά, οπότε αν χρειάζεται μετάφραση. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες και όλους. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και βέβαια να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερω την Επίτροπο Γιούροβα που παρίσταται στι εργασίε της ε, Επιτροπής μας απόψε, ε, απόψε. Πρώτο σημείο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν συμφωνείτε όλοι, να σας πω απλά ότι αν ολοκληρωθεί το επόμενο σημείο, δηλαδή η συζήτηση με την κυρία Γιώργα πριν τη ΣΕΝΕ, οπότε και προβλέπεται η ψηφοφορία, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε νωρίτερα και τις εκθέσεις για την απαλλαγή. Θα δούμε όμως ε, πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Δεύτερο σημείο της Μερσιάς Διάταξης, ανακοινώσεις της Προέδρου. έχετε λάβει αλλά έχει και αντίτυπα στο πίσω μέρος της αίθουσας μια μελέτη από το Ινστιτούτο των Φίλων για την ισότητα των δύο φίλων σε ό,τι αφορά την ε, διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Ελπίζω να είναι χρήσιμο το έγγραφο. Επαναλαμβάνω υπάρχουν αντίτυπα και στην αίθουσα αν θέλετε να τα πάρετε στα γραφεία σας. Οπότε περνάμε στο σημείο 3 της διάταξης όπου όπως σας είπα Καλωσορίζουμε την Επίτροπο, την κυρία Γιούροβα. η οποία θα συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Θα μιλήσει πρώτα η Επίτροπος, θα μας αναφέρει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ισότητας των φύλων. Εν συνεχεία θα έχουμε έναν πρώτο γύρο παρεμβάσεων θα μιλήσουν οι συντονίστριες των πολιτικών ομάδων καταρχάς. Θα απαντήσει η κυρία Γιούροβα και αν έχουμε χρόνο ενδέχεται να υπάρξει και ένας δεύτερος γύρος παρεμβάσεων από τους υπόλοιπους συναδέλφους, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το χρόνο, διότι η κυρία Γιούροβα θα πρέπει να μεταβεί στην Ολομέλεια. Οπότε μόνο αν υπάρχει χρόνος θα γίνει δεύτερος γύρος παρεμβάσεων. Τρία λεπτά θα είναι ο χρόνος των παρεμβάσεων για να υπάρξει δυνατότητα και ενός δεύτερου γύρου. Εδώ ολοκληρώνω και δίνω το λόγο στην Επίτροπο την κυρία Γιούροβα. Ευχαριστώ κύριε βουλευτές. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ για να συνεχίσουμε τον ε, δομημένο διάλογό μας ε, καθώς ε, αυτή είναι μια ευκαιρία για εμάς να εξετάσουμε την πρόοδο. Την πρόοδο που κάναμε το 2015 θα εξετάσουμε σήμερα λοιπόν και τα σχέδια για το 2016. Θα ζητήσω όμως συγγνώμη γιατί θα είμαι ε, βιαστική καθώς ε, πρέπει να πάω στην Ολομέλεια να αντικαταστήσω το, το συνάδελφο που ασθένησε. Δεν ήταν στο πρόγραμμα αρχικά αυτό. Να σας ε, παρουσιάσω τη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2015-2019 που εκδόθηκε στις 3 Δεκεμβρίου και αποτελεί το πλαίσιο για τη μελλοντική δουλειά της Επιτροπής για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων κατά τη διάρκεια της θητείας της μέχρι το 2019. Θα είμαι ξεκάθαρη, η Κομισιό παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην προώθηση της ισότητας των φύλων όπως ορίζεται στο πρόγραμμα του 2016 η στρατηγική είναι στην ουσία η συνέχεια, το follow-up της τρέχουσας στρατηγικής της ε, Κομισιόν για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 2010-2015. Ξέρω ότι πολλοί από εσά ανησυχείτε για την κατάσταση του εγγράφου και θα θέλατε μία ανακοίνωση που προσυπογράφει το Κολέγιο των Επιτρόπων. Όμως, η, ε, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν σημαίνει αυτό πως η ισότητα των φύλων έχει υποβαθμιστεί και έχει γίνει γίνει λιγότερο σημαντική. Είμαι το ίδιο παθιασμένη με αυτό το θέμα όπως και εσείς. Και εγώ επικεντρώνομαι στο περιεχόμενο. Στην καριέρα μου έχω δει πάρα πολλές στρατηγικές με πολλές λέξεις και λίγες δράσεις, λίγες πράξεις και λίγη πρόοδο δεν έχει νόημα ε, για την ε, ισότητα των φύλων αν ε, οι συζητήσεις σας μπουν σε ανακοίνωση ή σε έγγραφα εργασία. Για μένα είναι ευπρόσδεκτες στη στρατηγική 2010-2015 δράσεων που παραμένουν ενισχύ σήμερα. Η αξιολόγηση που κάναμε κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα μηνών και με τη δική σας συμβολή στην ουσία επιβεβαιώνουν όλα αυτά. Γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτούς τους τομείς προτεραιότητας που έχουν ε, ε, συνάφεια και με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ε, Ισότητα των Φύλων που συνεχίζει μέχρι το 2020. Η στρατηγική λοιπόν έχει τέσσερις θεματικές προτεραιότητες. Την αύξηση στη συμμετοχή, τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τη μείωση το διαφοράς τους μισθούς και τις αμοιβέ, την προώθηση της ισότητας ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, στην λήψη αποφάσεων και τέταρτον ε, πάταξη της βίας, υποστήριξη των θυμάτων και πέμπτον υποστήριξη της ισότητας των φίλων σε όλο τον κόσμο. Στη στρατηγική θέσαμε στόχους για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς και έχουμε και πιο συγκεκριμένες ε, δράσεις, 30 στον αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι επίτροποι έχουν δεσμευτεί για αυτή τη στρατηγική η οποία ορίζει το mainstreaming ως ε, μια γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το gender mainstreaming, και ε, δηλαδή την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και θέλουμε αυτό το πράγμα να μπει σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης. Με τους δείκτες λοιπόν και τα στοιχεία η στρατηγική προσπαθεί να δει πώς θα μετρήσουμε στο μέλλον την πρόοδο στον τομέα της οικονομικής ανεξαρτησίας με ίσους όρους για άντρες και γυναίκες μιλάμε για την συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση και το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το θέμα των ισορροπιών στην ε, εργασιακή ε, ζωή και έχουμε κάνει μια αξιολόγηση της οδηγίας ε, για την κοινωνική ασφάλιση, την πρόθεση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και θα αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες γυναίκες κατά την ε, και κατά την συμμετοχή τους στην αγορά ε, ε, εργασίας. Προσπαθούμε λοιπόν, μετά από αυτή τουλάχιστον την ανταλλαγή απόψεων, θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία για να μπορέσουμε να έχουμε μία, ένα σχέδιο με τους Τίμερμανς, τον και Τάισεν θα έχουμε συνεργασία ώστε ε, να ληφθεί μια νέα πρωτοβουλία για ένα νέο ισχυρό φιλόδοξο πακέτο ε, όσον αφορά στις άδειες μητρότητας, πατρότητας, ε, γονικές ε, και, φρο... και... κηδεμόνος. Επίσης θέλουμε να έχουμε και ευέλικτους χρόνους εργασίας και μια καλή πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες φροντίδας και την ε, σωστή ε, διανομή ας πούμε, των ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και ισότητα των φίλων σε κάθε παρόμοιο θέμα. Επίσης θα ήθελα να σας καλέσω να συμμετάσχετε σε μια διαβούλευση που θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου του χρόνου για τα θέματα αυτά. Θέλουμε να εργαστούμε σκληρά ώστε ήδη το 2016 να έχουμε αποτελέσματα και γι' αυτό θέλω να ακούσω από εσά τις απόψεις σας για αυτό το σημαντικό πακέτο προτάσεων για την οικονομική ανεξαρτησία. Όσον αφορά στην οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, αυτός ο, τομής, ο τομέας ε, έχει να κάνει με την ισότητα στη λήψη αποφάσεων. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε την έγκριση της πρότασης του 2012 για μια οδηγία που θα βελτιώνει την ισότητα των φύλων σε, όσον αφορά στα εκτελεστικά μέλη ε, εισηγμένων εταιριών. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη σε στοχευμένες πρωτοβουλίες που θα βελτιώνουν ε, την ε, ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων ε, όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων όπως, σε τομείς όπως η πολιτική, η έρευνα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά εντός του Κολεγίου των Επιτρόπων και με τις υπηρεσίες των Επιτρόπων. Θέλουμε λοιπόν να συμπληρώσουμε τα στοιχεία, λέξουμε και να μοιράσουμε στοιχεία που έχουμε συλλέξει σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Εξαιτία βέβαια τη αντίσταση 10 κρατών μελών δεν μπορέσαμε να πετύχουμε την ε, γενική προσέγγιση ε, στο Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας. Και πραγματικά έχω απογοητευτεί που δεν υπήρξε πρόοδο σε αυτό το θέμα παρά τις βαλτιστές προσπάθειες της Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη έχουν είχαν τον κατάλληλο χρόνο, αντιμετωπίσαμε τα θέματα της επικουρικότητας, δώσαμε την κατάλληλη ευελιξία ώστε να έχουν αποτελεσματικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Ήμουν ξεκάθαρη. Είπα ότι αυτή τη σημαντική πρόταση δεν θα την αφήσω να δηληστεί και τελικά ε, να πω ότι αυτή είναι μια προτεραιότητα για μας, ε, ε, ότι παραμένει προτεραιότητα και για το πρόγραμμα του 2016 και θα κάνω ό,τι μπορώ για την επιτυχία του. Επιπλέον, ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τα προβλήματα που αφορούν στις συντάξεις, ε, τις αμοιβέ και τους μισθούς ε, και έχουν να κάνουν ε, πολύ με τα προβλήματα που υπάρχουν γενικότερα στην αγορά εργασίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ε, αξιολογούμε την ε, οδηγία για την ίση μεταχείριση, την απασχόληση και ε, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις εταιρείες μέσα από τις πλατφόρμες για την ποικιλομορφία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που ξεκίνησε το 2014 και το οποίο ε, μια σύσταση την οποία αξιολογούμε αυτή τη στιγμή ε, θα μπορούμε να συζητήσουμε για τα συμπεράσματα. Θέλουμε η ισότητα των φύλων επίσης να προωθηθεί σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης αλλά και να προωθήσουμε και την απασχόληση γυναικών στο τομέα της, των ε, ΤΠΕ και σε κάθε μορφή υπηρεσιών. Σε συνεργασία με την κυρία Τάισεν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του χάσματος της συντάξης, της ανισότητας δηλαδή και θέλουμε να δημιουργηθεί ένας δείκτης ώστε να γίνεται μέτρηση και παρακολούθηση αυτών των στοιχείων. Μίλησα επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεχή προτεραιότητά μας όσον αφορά στην πάταξη της βίας λόγω φίλου ή ε, Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε με την διαθεσιμότητα των ε, στοιχείων ε, και την ε, ευαισθητοποίηση να έχουμε αποτελέσματα. Το 2016 θα πάμε στη... Θα συμμετάσχουμε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Επίσης θα υποστηρίξουμε την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων και θα συνεργαστούμε με τη Γύρωστατ και την ΕΓΚΕ στους δικούς τους τομείς δράσης. Επίσης θα υποστηρίξουμε την βάση δεδομένων για τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών και ε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι γίνεται για να πατάξουμε τον ακροτηριασμό και άλλες παρόμοιες ε, πρακτικές. Η ισότητα των φύλων είναι ένα θέμα που ε, υπάρχει και στην ατζέντα του 2013 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουμε συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό θα το κάνουμε μέσω δράσεων που ε, έχουν ήδη εισαχθεί μέσα στα πλαίσια των δράσεων για τις εξωτερικές ε, ε, την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργασία με την κυρία Μαργκερίνη προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό άμεσα. Να καταλήξω λέγοντας κάποια πράγματα για τη χρηματοδότηση. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθούν κονδύλια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική μας αποτελεί... Ε, έχει ε, μια χρωματοδότηση της τάξης των 6,17 δις για την περίοδο 2014-2020. Είμαι σίγουρη ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια σημαντική βάση για τις δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων τα επόμενα χρόνια και θα καλυφθούν όλα τα βασικά ζητήματα που έθεσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τον Ιούνιο του 2015. Η Προεδρία επίσης επιβεβαίωσε το στόχο της να εγκρίνει τις ε, προτεραιότητες ε, της Κομισιόν για το θέμα αυτό μέσα στο επόμενο ημίση του έτους. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε μεταξύ μας ε, πώς ακριβώς θα σχεδιάσουμε αυτό το εργαλείο, πώς θα έχουμε καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, πώς θα δράσουμε όσον αφορά στη σύμβαση της και πώς θα πιέσουμε για την ισότητα των φύλων στη λήψη αποφάσεων. Βασίζομαι σε εσά στη συνεχή συνεργασία σας και ε, αδιμονό, ώστε να συνεργαστούμε, να συνεργαστούμε στενά στο μέλλον ώστε να βελτιώσουμε την ισότητα των φύλων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιούροβα. Όπως είπα και στην αρχή, θα ακολουθήσει τώρα ένας γύρος παρεμβάσεων όπου θα λάβουν το λόγο οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Και έχουμε περιορισμό χρόνου. Τρία λεπτά ο κάθε ομιλητής. Αν υπάρξει χρόνος θα έχουμε και ένα δεύτερο γύρο όπου θα μπορούν να πάρουν το λόγο οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Κυρία Λεγκρίπ, εκ μέρους του ΕΛΚ, είναι η πρώτη μιλήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε και πρώτη το λόγο ως συντονίστρια από την ομάδα του ΕΛΚΑ. Θα ήθελα να μην εξαντλήσω τα τρία λεπτά ή δυνατόν για να δώσω τον λόγο σε άλλα μέλη της ομάδας μου. Κατάλαβα ότι δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή της και η Επίτροπος. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη για να ακούσουμε διάφορες απόψεις. Πρώτα απ' όλα να σημειώσω την προσήλωση, τη δέσμευση της Επιτρόπου μεταξύ άλλων ε, στα ζητήματα που άπτονται και της Επιτροπής Γυναικών. Σίγουρα έγινε πολλή δουλειά και από την αρχή της κοινοβουλευτικής αυτής ε, θητείας ε, και τους προηγούμενους ε, μήνες και σίγουρα ε, και εμείς έχουμε ενθαρρύνει και στηρίξει την ε, Επίτροπο αλλά και όλους τους άλλους επιτρόπους που είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουν να δηλώνουν το παρόν και να τα αποκρίνονται στις προσδοκίες και τις δικές μας και όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Για λόγους ίσως ε, υπερβολικής τυπολατρείας ή καθυστέρηση ε, για τη διαδικασία λήψη ε, αποφάσεων εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ήταν δυνατόν Ίσως για αυτούς τους λόγους να έχουμε ακριβώς το ίδιο είδος εγγράφου που είχαμε την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Όμως το σημαντικό είναι όχι τόσο ο τύπος αλλά η ουσία. Το Engagement for Gender Equality αυτό το έγγραφο λοιπόν για την περίοδο 2016-2020 έχει ε, πολλά κεφάλαια και συγκεκριμένες ε, δεσμεύσεις. Αυτή η γραμμή λοιπόν που θα ακολουθηθεί τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια θέλουμε ο ΣΕΛΚ να είναι συγκεκριμένη και να έχει στόχο την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων και να ε, μπορεί ε, να στηρίξει και τα κράτη-μέλη και να τα οθήσει να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να παίξετε κι εσείς αυτό το ρόλο ενθαρρύνοντας και προ, ε, παροτρύνοντας τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Η ε, Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κυρία Λεγκρίπ, εκ μέρους Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Αρενά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την παρουσίασή σας αυτή. Δεν θα σας κάνει εντύπωση όταν λέω ότι δεν συμφωνώ με την Constance Legri όσον αφορά το ζήτημα της, του τύπου του καθεστώτος του εγγράφου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί η ανακοίνωση δίνει διαφορετικό καθεστώς στη στρατηγική που μας περιγράψατε. Και μπορούμε μέσω του καθεστώτος αυτού με το σύνολο των επιτρόπων να έχουμε μια κοινή στρατηγική. Τη στρατηγική μας περιγράψατε. Δεν θα πρέπει δηλαδή η στρατηγική αυτή να εμπίπτει μόνο στη δική σας αρμοδιότητα όπως είπατε, είναι και η Επίτροπος η για την απασχόληση. Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε και με άλλες πτυχές, όπως η χρηματοδότηση, η ειδική χρηματοδότηση για τις πολιτικές ισότητας των φύλων. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές πτυχές που εμπίπτουν η στρατηγική αυτή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε πραγματική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε προκειμένου να καταλήξετε ως Επιτροπή σε πραγματικό κείμενο ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρετε να καταρτήσετε και μια πολιτική σε σχέση με τις προτεραιότητες που μας περιγράψατε. Θα μπορούσατε λοιπόν με τη βοήθεια τόσο του Συμβουλίου όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταλήξετε στο κείμενο αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, σε ένα πρόσφατο συμβούλιο τα ίδια τα κράτη-μέλη είπαν ότι θέλαν και αυτά να καταλήξετε εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια επίσημη ανακοίνωση. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού, ομολογώ ότι εγώ θα ξεκινούσα από την πρώτη προτεραιότητα που είναι η βία κατά των γυναικών. Φαινόμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα υπαρκτό ακόμα. Είπατε ότι προσωπικά δεσμεύεστε για την πάταξη της βίας κατά των γυναικών. Έχει περάσει όμως ένας χρόνος από τότε που αναλάβατε τη δέσμευση αυτή και ακόμα μιλάμε για το αν τελικά θα εφαρμοστεί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Το 2016, 2017, 2018, 2019 θα λέμε ότι προτιθέμεθα να επικυρώσουμε τη σύμβαση αυτή χωρίς όμως να το πράττουμε στην πράξη. Τι γίνεται λοιπόν με την περίφημη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ζήτημα το οποίο συνδέεται και με τις γυναίκες μετανάστες και τη βία που δέχονται πολλές φορές οι γυναίκες αυτές και αναφέρομαι προφανώς επίσης και στις γυναίκες οι οποίες κάνουν αίτηση για άσυλο και πολλές φορές καθ' όλη τη διάρκεια της μεταστατικής διαδικασίας υφίστανται φαινόμενα βία. Βίας. Όσον αφορά τώρα τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ε, ζωής. Ξέρετε ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οδηγία για την γονική άδεια και την άδεια μητρότητας. Δυστυχώς τελευταία κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας είπα ότι θα επανέλθετε με κάτι το πιο σύγχρονο. Αν όμως οι κοινωνικοί εταίροι και ιδίω οι εργοδότε είναι κατά της γονικής άδειας, τι προτίθεστε εσείς να κάνετε. Πρόκειται για μια οδηγία που υποστηρίζεται από του κοινωνικού εταίρου. Εσεί, αν δεν συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, θα υποβάλλετε μια πρόταση οδηγία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αφήσω τι συναδέλφου να πάρουν το λόγο για τα υπόλοιπα σημεία. Να αναφερθώ προς το ζήτημα των δικτών. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σωματώσουμε του δείκτε τη ισότητα των φύλων σε όλε τι πολιτικέ παρακολούθησει που έχουμε, ακόμα και στα πλαίσια τη ανάλυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, διότι ξέρετε ότι οι πολιτικέ λιτότητα βάλουν ιδίω κατά των γυναικών. Πρέπει λοιπόν να σωματώσουμε και τέτοιου δείκτε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κυρία Αρενά, εκ μέρου τη ομάδα Άλντε, η κυρία Μπέρντερ. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο που είναι σήμερα μαζί μας και μας δίνει και μία ε, ενημέρωση για τη δουλειά της. Έχω δύο σύντομες ε, ερωτήσεις γιατί θα ήθελα και εγώ να δώσω χρόνο στη συναδελφό μου. Ε, σε συνέχεια του ό,τι είπε και η συνάδελφος Καρίνα για την ισορροπία μεταξύ της ιδιωτικής και της ε, επαγγελματικής ζωής, θα ήθελα να υπογραμμίσω την θετική διάσταση της δουλειάς της Κομισιόν σε αυτό το θέμα. Ήσασταν πραγματικά πολύ ενεργή σε προληπτικό επίπεδο και ήθελα να ρωτήσω τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν σε αυτό το επίπεδο, τι είναι καινούριο. Ποια είναι η στρατηγική της Κομισιόν για να μπορέσει να ξεπεράσει το διέξοδο αυτή τη φορά στο Συμβούλιο. Δεύτερον, η ερώτησή μου έχει να κάνει ε, με τις πρωτοβουλίες για την προώθηση των ε, δικαιωμάτων ε, των ε, ΛΟΑΔΜ. Ήθελα να ρωτήσω τι θα κάνει η Κομισιόν, η Ολλανδική κυβέρνηση έχει πραγματικά δεσμευτεί ότι θα αναλευθούν πραγματικές πολιτικές ευθύνες για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε κυρία Μίλνερ. Μέρος της Γκουε τώρα. Η κυρία Πιόρκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, που, κυρία Επίτροπε που είστε εδώ για έναν ε, επικοδομητικό διάλογο. Ε, ανησυχούμε όπως είπα την υποβάθμιση ε, του εγγράφου. Είναι ένα εγγραφό εργασίας και πραγματικά χρειαζόμαστε πολιτικά ε, έγγραφα που να μπορούν να οδηγήσουν σε πολιτικές ε, λύσεις. Δεν χρειαζόμαστε έγγραφα εργασίες. Εδώ ασχολούμαστε με τον φεμινισμό, τις γυναίκες. Είμαστε καθημερινά λοιπόν εδώ και με θάρρος εργαζόμαστε και δεν φτάνει ένα εγγραφό εργασίας. Χρειαζόμαστε έγγραφα πολιτικής καθοδήγησης γιατί αυτός ο αγώνας που δίνουμε και για τα δικαιώματα ψήφου και για τα σωματικά μας δικαιώματα ως γυναίκες είναι πράγματα που ε, πρέπει να αναγνωριστούν μέσα από αυτό το μήνυμα που θα σταλεί από ένα τέτοιο έγγραφο. Όπως ήδη υπόθηκε, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν στο έγγραφο. Θα επανέλθω ε, να και θα πω ότι πρέπει να υπάρχουν ε, νομοθετικές προτάσεις για τη βία κατά των γυναικών ε, και πραγματικά ε, θα ήθελα να υπήρχε και μια νέα σύμπραξη μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για αυτό το θέμα. Θέλουμε πολιτική ισχύ και ηγεσία για τα project που έχουμε. Γιατί αλλιώ ε, θα απογοητεύσουμε όλους, όλες τις φεμινίστρες και τις γυναίκες που εργάζονται σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ κύριε Πιόρκ. Κυρία Ρέντκε από τους Πρασίνους τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και προσωπικά και η ομάδα μου θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε κυρία Γιούρουβα για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολος ο αγώνας που δίνεται στο Σώμα των Επιτρόπων κυρία Γιούρουβα για την ε, ισότητα των φίλων. Και πρέπει να σας πω ότι και εμείς πράγματι απογοητευθήκαμε βλέποντας ότι αυτό που μας παρουσιάζεται είναι ένα έγγραφο εργασίας απλά. Αυτό μας απογοητεύει. Φαντάζομαι και εσείς θα θέλατε κάτι διαφορετικό. Ήθελα να το πω όμως. Δεν πρόκειται για ρεαλισμό ε, ή το ότι θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα σημεία. Όλοι το θέλουμε αυτό και δεν θέλουμε μακροσκελή έγγραφα. Θα περιστώ σε τέσσερα σχόλια και θα σας παρακαλέσω να μας δώσετε γνήσιες ειλικρινές απαντήσεις. Πρώτον, είπατε σαφή νομοθετικά μέτρα για την γονική άδεια, την άδεια μητρότητα, την άδεια πατρότητα. Θα υπάρξουν νομοθετικές προτάσεις. Επειδή αποσύρθηκε η οδηγία για την άδεια μητρότητας και σε ό,τι αφορά τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, ξέρω ότι αγωνίζεστε να περάσει αυτή η πρόταση στο Συμβούλιο όμως για ιδεολογικούς λόγους κάποια κράτη-μέλη μπλοκάρουν αυτή την πρόταση. Και τι θα πει ε, ότι μπορεί να ε, γίνει μια προσπάθεια να σκεφτούν πιέσεις ε, επί Ολλανδικής Προεδρίας. δεύτερο θέμα, βία κατά των γυναικών. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης προσχώρησε αυτή τη σύμβαση, είναι σημαντικό. Αλλά δεν έχουμε σε ό,τι αφορά τη βία των γυναικών στο ενωσιακό δίκαιο κάποια ε, διατάξεις. Είχαμε ακούσει κάποιες ε, φήμες βέβαια. Επίσης αναφέρατε το ρόλο των γυναικών στο ψηφιακό θεματολόγιο. Θα γνωρίζετε ίσως ότι έχουμε έκθεση πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή. Και εστιάζω μεταξύ άλλων ήταν και μια προτεραιότητα άλλωστε που ανέκυψε από τη συζήτηση, είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για γυναίκες επιχειρηματίες και γενικά για την πρόσβαση των γυναικών ε, σε χρηματοδότηση στο ψηφιακό τομέα. Μιλήσατε για χρηματοδότηση. Έχουμε το ψηφιακό θεματολόγιο, οι πόροι που διατίθεται στο πλαίσιο του θεματολογίου αυτού ή τέλο πάντων κάποιο μέρο αυτών των χρημάτων θα μπορούσαν να δοθούν ε, σε γυναίκε ή για γυναίκε. Αν δεν υπάρχουν στοχευμένα ε, προγράμματα, οι γυναίκε έχουν πολύ λιγότερη πρόσβαση σε τέτοιου είδου κονδύλια. Αν θέλουμε όμω ε, να συμμετέχουν στο λογοψηφιακό θεματολόγιο οι γυναίκε, θα πρέπει να του εξασφαλίσουμε αυτή τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέντκη. Η κυρία Γιούτα από το FND. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε. Λυπάμαι που δεν κατάφερα να ακούσω όλη την παρουσίασή σας. Πάντως πιστεύω ότι τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Πρέπει να δούμε επίσης πώς διαμορφώνεται το φαινόμενο αυτό στην παρούσα συγκυρία, στην κυρία της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Ξέρετε ότι το φαινόμενο αυτό έχει ενταθεί Ζούμε επίση σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τρομοκρατικέ επιθέσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, μόνο και μόνο η ε, παρουσία όλων αυτών των φαινομένων, ο συνδυασμός επίσης ε, Ισλαμισμού και οι γυναίκε είναι κάτι το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει περισσότερο. Η θέση των γυναικών δηλαδή στο νέο αυτό περιβάλλον που διαμορφώνεται, που είναι αρνητικό για τις γυναίκες. Έπειτα, τα κίνητρα τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν για να έχουμε περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Προφανώς ξέρετε ότι εμείς θα μπορούσαμε να χαιρετήσουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση των γυναικών σε τέτοια διοικητικά συμβούλια. Ωστόσο, δεν είμαστε υπέρ των ποσοστώσεων για τις γυναίκες. Είμαστε πεπισμένοι ότι άλλα μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Να χρησιμοποιηθούν. Θα πρέπει για παράδειγμα να ενισχυθεί και ε, η κοινωνική κατάσταση όσον αφορά τις γυναίκες και η κοινωνική πρόνοια, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας για τις γυναίκες. Ως προς αυτό, ποια μέτρα προτίθεστε εσείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνετε υπέρ των γυναικών. Προβλέπετε μια κάποια ενίσχυση του συστήματος αυτού, του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας για τις γυναίκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γιούτο. Εδώ ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος. Ακούσαμε τις παρεμβάσεις των συντονιστών, συντονιστριών καλύτερα. Κύριε Γιούροβα, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Yes, thank you. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. I will try to reply. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες ε, μέσα στο χρονικό διάστημα που έχουμε. Καταρχάς θα ήθελα να μιλήσω για το νομικό ε, καθεστώς ε, και την μορφή, τον τύπο τη στρατηγική. Πριν από αρκετό καιρό ήμουνα σε μία ακρόαση, δεν ήταν και ωραία τότε, μπορώ να πω, και με ρώτησαν για τη στρατηγική και είπα ναι, θα φέρω τη στρατηγική εν ευθέτω χρόνο και θα περιλαμβάνει τους βασικούς στόχους, τις προτεραιότητες, τις δράσεις, τους μετρήσιμους δείκτες, τη χρηματοδότηση και τους όρους χρηματοδότησης, και τον ορισμό των ε, αρμόδιων φορέων. Και αυτό έκανα. Ε, οπότε νομίζω είναι ε, μια μικρή παρεξήγηση αυτό που έχει γίνει η δέσμευση για τη στρατηγική. Είναι στην ουσία μια πραγματική στρατηγική, ένα εργαλείο σχεδιασμού για την Κομισιόν και για άλλους που μπορούν να συνταχθούν με μας και να εργαστούν στον τομέα της ισότητας των φύλων. Σας κατανοώ ε, και κατανοώ και τους ε, υπουργούς όταν με επέκριναν ε, πολύ την περασμένη εβδομάδα, τη Δευτέρα, και στην ουσία είπαν ότι πρόκειται μόνο για ένα έγγραφο εργασίας όμως εγώ προσωπικά ε, δεν θεωρώ ότι αυτές οι ανησυχίες επηρεάζουν στην ουσία την αποτελεσματικότητα του εγγράφου. Γιατί ε, χρειάζεται να προχωρήσουμε και να το κάνουμε. Να κάνουμε αυτά που έχει μέσα του το έγγραφο, το περιεχόμενό του να το εφαρμόσουμε. Άρα εκτιμώ τις επικρίσεις σας, ίσως αν ήμουν και εγώ στη θέση σας να επέκρινα κι εγώ γιατί είναι τόσο προφανές ότι έχουμε τώρα ένα έγγραφο με διαφορετικό νομικό καθεστώς όμως αν το συγκρίνουμε με την προηγούμενη στρατηγική και δεν θέλω να επικρίνω τους ε, προκατόχους μου και τους ε, συναδέλφους μου τους τωρινούς όμως η προηγούμενη στρατηγική δεν είχε ε, ξεκάθαρα απτούς στόχους που μπορούσαν να μετρηθούν. Αυτό το έγγραφο λοιπόν που πήραμε στα χέρια μας και, όταν και θελήσαμε να δούμε τι δούλεψε και τι δεν δούλεψε και ποια ήταν τα αποτελέσματα, συνειδητοποίησαμε ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε αυτές τις πληροφορίες, γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ γενικό και οι μετρήσιμοι στόχοι δεν είχαν οριστεί ξεκάθαρα. Για να ορίσουμε στόχους μετρήσιμους και να δεσμευτούμε ως προς αυτούς, πρέπει να έχουμε και κάποια λογοδοσία. Είμαι λοιπόν έτοιμη να λογοδοτήσω για αυτά που κάνω στην πολιτική της ισότητας των φίλων. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, πραγματικά δεν είναι εύκολη η δουλειά μου, όντας ε, η Επίτροπος υπεύθυνη για την ισότητα των φίλων εντός του κολεγίου. Ε, το πιο εύκολο κομμάτι της δουλειάς μου είναι εδώ, να πω. Γιατί εδώ με υποστηρίζετε. Υποστηρίζετε τις ιδέες για την ισότητα των φύλων και προχωρούμε και προωθούμε και σπρώχνουμε όλους τους συναδέλφους που δουλεύουν για την καλύτερη συμμετοχή σε αυτό το θέμα της ε, ισότητας των φίλων. Να πω λοιπόν ότι μάχομαι εντό της Επιτροπής ε, ε, και αυτή η στρατηγική ήταν αποτέλεσμα πολύ σημαντικών διαβουλεύσεων και δεσμεύσεων που μπόρεσαν οι συνάδελφοι επίτροποι να λάβουν από τη δική τους πλευρά, είτε πρόκειται για τον Επίτροπο Υγείας, Περιβάλλοντος ή Μεταφορών. Πρόκειται για μια ισχυρή δέσμευση λοιπόν από την πλευρά της Επιτροπής και είμαι περίεργη να δω και την αντίδραση των κρατών μελών όταν ε, την επόμενη άνοιξη θα πρέπει να αποφανθούν γιατί έχω ζητήσει από αυτούς να παίξουν και αυτοί το δικό τους ρόλο και να συνδέσουν τις στρατηγικές και τα σχέδιά τους με τη δική μας δέσμευση για τη στρατηγική, έτσι ώστε να έχουμε πραγματική πρόοδο και αποτελέσματα στο πεδίο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να κάνετε το ίδιο, γιατί θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο περιεχόμενο. Αν ε, με επικρίνετε πολύ ε, αυστηρά λέγοντας ότι δεν έχω κάνει αρκετά κατά της βίας των, ε, κατά των γυναικών, για μένα αυτό αποτελεί μια όθηση ώστε να το κάνω καλύτερα και με μεγαλύτερη στεναρότητα αυτό που κάνω. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα, σχέδια, δράσεις που δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω της νομοθεσίας. Αυτά πρέπει να πετύχουμε με εντατική εργασία μη, νομοθετικού, μη νομοθετικής φύσεως στα κράτη-μέλη και γι' αυτό θέλω σήμερα να σας ζητήσω την συνεργασία σας και σε αυτόν τον τομέα γιατί χρειάζεται μια ε, σημαντική εκστρατεία, προσωπικά παραδείγματα ή, ή, φωνές που θα ακουστούν. Και θα μιλώντας για την βία κατά των γυναικών και άλλα τέτοια φρικτά πράγματα. Για να απαντήσω τώρα και τις άλλες ερωτήσεις. Ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Θα είμαι συγκεκριμένη. Ναι, έχουμε λοιπόν νομοθετικές προτάσεις, τις οποίες θα έχουμε όταν λάβουμε τα αποτελέσματα από τους κοινωνικούς εταίρους, από τη διαβούλευση δηλαδή. την Τετάρτη Ιανουαρίου θα έχουμε λάβει τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και ε, έχουμε ήδη κάποιες προτάσεις στο τραπέζι μας, πολύ καλές, που τις έχουμε δουλέψει με τη Γενική Διεύθυνση. Οπότε τότε θα είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε άμεσα να έχουμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους συγκεκριμένες προτάσεις. Θα είναι μείγμα, το κάνει η Κομισιόν, νομιοθετικών προτάσεων που θα είτε ενημερώνουν, για να το πω καλύτερα, ή τέλο πάντων θα αντικαθιστούν την οδηγία για την μητρότητα όσον αφορά στο θέμα των διαφόρων αδειών, μητρότητας, πατρότητας κτλ. Η οδηγία για την άδεια μητρότητα είναι παλιωμοδίτικη. Δεν οδηγεί τους άντρες στη συνεργασία, δεν τους κάνει δηλαδή να βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού, στο νοικοκυριό. Και το δικαίωμα της μητρότητας δεν είναι το μοναδικό στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε στη ζωή γενικότερα. Αυτά που τώρα λέω όμως γενικά θα σας τα πω αργότερα πολύ πιο συγκεκριμένα όταν θα έχουμε και τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων. Something uh, επίσης στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και στην βία κατά των γυναικών. Για μένα θα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δυνηρό τμήμα της πολιτικής για την ισότητα των φύλων. Έχουμε δύο βασικά καθήκοντα εδώ πέρα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να ενισχύσουμε τη θέση των γυναικών. Ουσιαστικά θα πρέπει να προσφέρουμε καταρχάς για τις πιο ισχυρές δυνατές γυναίκες συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού και δεύτερον θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις πιο αδύναμες γυναίκες μελετήσαμε διάφορα δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν ότι ε, η βία συνδέεται άμεσα με την οικονομική ε, αδυναμία. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση στο φαινόμενο και να εξαντλήσουμε όλα τα στάδια τα οποία πρέπει να εξαντλήσουμε προκειμένου να μειώσουμε και το μισθολογικό χάσμα και να πολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών. Στην πράξη πώς μπορεί να γίνει αυτό. Η προσχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη Σύμβασης Κωνσταντινούπολης ενέχει μια νομοθετική διαδικασία. Θα πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να τιμωρήσουν αυτό το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, να προβλέψουν οι κυρώσεις. Πρόκειται για ένα ποινικό αδίκημα άλλωστε και πρέπει παράλληλα να χρησιμοποιήσουμε σωστά όλα τα διαθέσιμα κονδύλια προκειμένου να προωθήσουμε όλους τους μη κυβερνητικού οργανισμούς που ειδικεύονται στην καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε στην πράξη τις γυναίκες που είναι θύματα αυτού του φαινομένου. Όσον αφορά τώρα την νομοθεσία, σας παραπέμπω στην οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων ένα 10 με 15% μόνο των γυναικών αυτή τη στιγμή καταγγέλουν ότι είναι θύματα της βίας λόγω φύλου, λόγω εξαιτία του γεγονότος ότι είναι γυναίκες και καταλαβαίνετε το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Θα πρέπει να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο, να προασπίσουμε περισσότερο τα δικαιώματα των θυμάτων. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε που φοβούνται να πάνε στην αστυνομία για να καταγγείλουν τα φαινόμενα αυτά, γιατί πολλοί αστυνομικοί ενδεχομένως και θα το πω μπορεί να συμπεριφερθούν εντελώς ε, ανόητα και να καταγγείλουν τελικά, ε, να αποδοκιμάσουν την ίδια τη γυναίκα, να πούνε στη γυναίκα ότι εσύ το προκάλεσες τελικά, ότι εσύ είσαι η υπεύθυνη για το φαινόμενο αυτό. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και ξέρουμε ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πήγαν στην αστυνομία και δυστυχώς εκεί πέρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με αυτό το εντελώ αρνητικό για αυτές περιβάλλον, με μια αντιεπαγγελματική στάση από πλευρά της αστυνομία. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι όντω οι γυναίκε θα την χάνουν τη σωστή συμπεριφορά κάθε φορά που καταγγέλνουν τέτοια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα τι ομάδε ΛΟΑΔΜΑ, η Ολλανδική Προεδρία υποσχέθηκε ότι θα κάνει κάθε τι το δυνατό προκειμένου να προωθήσει την έγκριση της οδηγίας για την ισότιμη μεταχείριση. Δεν είμαι ικανοποιημένη από την πορεία της οδηγίας αυτής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις, γιατί προβλέπεται στα πλαίσια της οδηγίας ότι θα μπορούν να προβλέπονται συγκεκριμένες νέες υποδομές για, για τα άτομα που έχουν ειδικέ ανάγκες και το πρόβλημα είναι ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν αρχίσει ήδη να καταμετρούν πόσο θα τους στοιχήσει η εφαρμογή μιας τέτοιας οδηγίας. Θα ήθελα λοιπόν μια πιο επικοδομητική προσέγγιση στην οδηγία αυτή από τα κράτη-μέλη σε κάθε περίπτωση η Ολλανδική Προεδρία ότι θα την προωθήσει. Επίσης θα έχουμε και μια συνδιάσκεψη στην Δανία στα πλαίσια της οποίας θα γίνει και μία ισχυρή εκστρατεία με τη βοήθεια της Ολλανδικής Προεδρίας για την ισότιμη μεταχείριση και θα έχουμε και μία συνεδρίαση υψηλόβαθμη για την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης και θα μπορέσουμε εκεί πέρα να κάνουμε μια επικοδομητική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών όσον αφορά την αντιμετώπιση της διακριτικής μεταχείρισης των ομάδων ΛΟΑΔΜΑ. Νομίζω ότι ήδη η Ολλανδία έχει μια πολύ τέτοια θετική εθνική πολιτική, επομένω μπορούμε να ακολουθήσουμε την ηγετική στάση που προτίθεται να δείξει. Πρέπει να αποχωρήσω όμω τώρα. Σα ευχαριστώ πολύ για τι παρατηρήσει και τι ερωτήσει σα και προσβλέπω σε μια θετική συνεργασία μαζί σα. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιούροβα. Βέβαια έχουμε ένα μακρύ κατάλογο ετούντων το λόγο. Αν λοιπόν η Επιτρόπος συμφωνεί, η Γραμματεία θα συλλέξει μία ερώτηση από κάθε έναν και κάθε μία συνάδελφο που δεν μπόρεσε να πάρει το λόγο σήμερα και θα σας τις αποστείλουμε. Οπότε θα μπορείτε να απαντήσετε γραπτώς σε αυτά τα ερωτήματα, διότι η συζήτηση αυτή τη στιγμή πρέπει να λήξει, καθότι η Επίτροπος ε, πρέπει να, να τα βρει στην Ολομέλεια, όπως ε, Διακόπτεται η πρόεδρος. Okay, uh, let's, let's I, I am not... Uh, <laughs> Κοιτάξτε, ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν χρονομετρούσα κιόλα. Αλλά είναι έκτακτη αυτή η κατάσταση. Μακάρι να μπορούσα να μείνω. Εγώ δεν είχα σχεδιάσει ε, να έχω κάποια άλλη συνεδρίαση ε, μετά από αυτήν, αλλά αντικαθιστώ ένα συνάδελφο που αρρώστησε η πρόεδρος. Τρεις συνάδελφοι θα λάβουν το λόγο, αλλά παρακαλώ να διατυπώσετε συγκεκριμένα ερωτήματα και να μην επαναλαμβάνονται ερωτήματα που έχουν διτεθεί στην Επιτροπή. Κύριε Πετήρ.

E, Κυρία Επίτροπε Γιούροβα, έχω μια ερώτηση για την οδηγία περί ισότιμης μεταχείρισης, μάλλον ισότητας ευκαιριών. Θα δεσμευτείτε προκειμένου να εστιάσει τον πρώτο τη στόχο αυτή η οδηγία, δηλαδή στα άτομα με αναπηρία. Διότι έχω την εντύπωση ότι δεν ακολουθούμε το σωστό δρόμο σε ό,τι αφορά τον ορισμό των διακρίσεων. Άρα παραβιάζονται πολιτικές αστικές ελευθερίες αλλά και η ιδιωτική ζωή των προσώπων. Και υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις και δυσαρέσκειες σε σχέση με αυτήν την οδηγία, ιδίω από τον ιδιωτικό τομέα. Δεσμεύεστε λοιπόν και επίτροπε να βοηθήσετε να δημιουργήσουμε ισότητα ευκαιριών με αυτήν την οδηγία για τα άτομα με αναπηρία και να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή διάκρισης. Στην οδηγία αναφέρονται διάφορες μορφές διάκρισης. Μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι το ίδιο ο σεξουαλικός προσανατολισμός ε, με την αναπηρία, για παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, τα τρία τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε όξυνση των ανισοτήτων και των διαφόρων. Και ιδίως ό,τι αφορά τα διοικητικά συμβούλια υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουμε καλύτερο εταιρικό πνεύμα και αύξηση του ΑΕΠ κτλ. Μήπως θα έπρεπε να ακούσουμε τους επιχειρηματίες γιατί δεν ε, είναι μόνο θέμα στρατηγικού, στρατηγικής σκέψης ή ε, ισολογισμοί, είναι και πώς ε, μεταφέρονται στην πράξη. Έχουμε κάποιες ποσοστώσεις για τα διοικητικά συμβούλια. Τι σκοπό έχουν αυτές τις ποσοστώσεις, να μπορούν να βρουν μια καλή θέση, μια καλή δουλειά γυναίκες. Και υποτίθεται ότι η Νορβηγία ήταν πρότυπο. Υπήρχε 40%. Το αποτέλεσμα όμως τελικά δεν ήταν και τόσο ικανοποιητικό. Διότι το 98% των γενικών διευθυντών παραμένουν άνδρες, κύριε Επίτροπε. Σε αυτά τα δελτα σίγμα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν γυναίκες, η διαδικασία δεν προχώρησε. Παρέμεινε στα <coughs> κατώτατα επίπεδα. Στη Λετωνία έχουμε πολλές γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια αλλά δεν επηρέαζαν τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, με αυτές τις ποσοστώσεις για την ε, παρουσία περισσότερων γυναικών ε, στα ανώτατα κλιμάκια. Τι προτάσεις θα κατεβάσετε για να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην ε, δίκηση των επιχειρήσεων. Κυρία Χάιντι. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ που είστε εδώ και από απαντάτε στις ερωτήσεις μας. Και εγώ πραγματικά απογοητεύτηκα όταν είδα ότι δεν είναι στρατηγική αλλά έγγραφο εργασίας αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι όπως υπόθηκε ήδη, νο, ε, είπαν, ήδη οι συναδελφοί, η νομική θέση ενός ε, εγγράφου εργασίας είναι διαφορετική. Όσον αφορά στη μάχη για τα δικαιώματα των γυναικών, είπατε ότι τη δίνετε και μεταξύ των συναδέλφων σας. Ε, σας καταλαβαίνουμε όμως συνεχώς οι γυναίκες και μάχονται ε, για τα ισότητά τους με τους άντρες, όχι μόνο εδώ, αλλά και εκτός ε, στην πραγματική ζωή και χάνουν ε, πάρα πολύ αν έχουν ένα έγγραφο εργασία απλώς. Πρέπει πραγματικά να καταλάβετε ότι υπάρχουν αμφιβολίες όταν κανείς για χρόνια παλεύει για τα δικαιώματα των γυναικών ε, για να υπάρχουν ε, ίσες αμοιβέ για την ίδια δουλειά και δεν πετυχαίνει όλα όσα θέλει, είναι απογοήτευση να έχουμε απλώς ένα τέτοιο έγγραφο. Είπατε ότι η παλιά στρατηγική ε, ήταν κακή, αλλά η απάντηση αυτή δεν αρκεί. Θα μπορούσατε να έχετε κάνει μια καλύτερη στρατηγική. Η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ ε, την ε, ε, Επιτροπή. Είμαστε όλοι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας εκπροσωπούν οι Επίτροποι. Οι Επίτροποι λοιπόν δεν εκπροσωπούν τα δικά τους κράτη-μέλη και όλα τα κράτη-μέλη εκπροσωπούνται ισότιμα στην Επιτροπή έτσι ώστε να ε, επιλύονται με τον ίδιο τρόπο και ισότιμα τα προβλήματα. Έχετε την αίσθηση ε, ότι υπάρχει αλληλεγγύη ε, ως προς τις γυναίκες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Υπάρχει δηλαδή αυτό το θέμα, υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ της Δυτικής και Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ε, ειδικά τώρα που εσείς είστε από την Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν τεράστιες ας πούμε διαφορές ε, στους μισθούς. Μια νοσοκόμα ε, παίρνει το ένα δέκατο στη, μια, χώρα, στη χώρα μου από την στην Αυστρία. Μια δασκάλα, κάποια γυναίκα που φροντίζει ε, ηλικιωμένους για παράδειγμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν αμείβονται το ίδιο ε, όπως οι άντρες. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να ε, διερευνήσουμε πιο βαθιά αυτό το ζήτημα. Βλέπετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες ε, από την Ουγγαρία για παράδειγμα ε, νοσοκόμες, ε, δασκάλες, ε, κοινωνικές λειτουργοί μεταναστεύουν από την Ουγγαρία προς τη Δυτική Ευρώπη. Υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρώπη γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα μου είναι το γεγονός ότι μας ανισχύει ιδιαίτερα πως οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Έχετε σκοπό να δείτε και να εξετάσετε ποια είναι η επιρροή αυτών των γυναικών στις αυτόχθονες γυναίκες. Γίνονται πιο βίες. Τι γίνεται. Ε, έχει πραγματικά αυξηθεί η βία. Έχει γίνει κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια έρευνα επίσης για την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων. Έχουμε τώρα και την παράνομη μετανάστευση. Ποια είναι η επιρροή που έχει μετανάστευση στις Ευρωπαίες γυναίκες. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Πώς γίνεται λοιπόν, ε, τι γίνεται λοιπόν με αυτό το θέμα, έχετε σκοπό να το διερευνήσετε. Κυρία Γιούροβα, έχετε το λόγο. Yes. Μάλιστα. Γρήγορα. Εκτός ε, μικροφώνου. Η πρόεδρος, ακούστε παρακαλώ. Εγώ προσπάθησα να δώσω το λόγο σε όλες τις συντονίστριες. Έπειτα έδωσα το λόγο στις ε, κεστούς, στην αδέλφους, ανάλογα με την ε, σειρά που είχαν σηκώσει το χέρι τους. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον έχουμε ολοκληρώσει και γι' αυτό πρέπει να απαντήσει η Επιτροπός. Λοιπόν, οδηγία για την ισότιμη μεταχείριση. Αυτή η οδηγία καλύπτει τα κενά της οδηγίας κατά των διακρίσεων. Από το 2008 νομίζω είναι αυτή η οδηγία. Δεν θα προβούμε σε κάποιες αλλαγές ε, στην παρούσα φάση, διότι όπου να θα εγκριθεί στο Συμβούλιο είναι στην ε, τελευταία φάση, ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις. Ε, νομίζω μια συντονίστρια έθεσε το ίδιο ερώτημα στον πρώτο γύρο. Εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε την οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι καταπληκτικοί και ικανότατοι άνδρες θα πρέπει να αντικατασταθούν από ανίκανες αναλφάβητες γυναίκες. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο η οδηγία, ούτε αυτό το σκοπό έχει. Αυτό που επιδιώκει είναι, όπως είπα, είναι να προωθήσει το δίκαιο ανταγωνισμό. Δηλαδή, οι υποψήφοι, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις απαιτήσει ό,τι αφορά τα τυπικά προσόντα, την εμπειρία, την παιδεία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και όταν είναι ισότιμοι οι υποψήφοι, να έχει προτεραιότητα το υποεκπροσωπούμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο φίλο. Περί αυτού πρόκειται. Θα μπορούσε να είναι και ο άνδρας που θα έχει προτεραιότητα αν στο Διοικητικό Συμβούλιο της δεδομένης εταιρείας είναι περισσότερες οι γυναίκες. Μπορεί να σας εκπλήξει αυτό βέβαια, αλλά τέτοιο Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Όσο έχει όμως τώρα η οδηγία, είναι ουδέτερη ως προς το φύλλο, διότι μιλά για υποεκπροσωπούμενο φύλλο. Το ότι ε, στην περίπτωση, μάλλον στις το 100%, στο 100% των περιπτώσεων ε, το υποεκπροσωπούμενο φύλλο είναι οι γυναίκες, αυτό κάτι λέει σίγουρα. Θέλουμε να φτάσουμε γύρω στο 30% και σίγουρα πρέπει να βρούμε περισσότερη υποστήριξη, διότι εξακολουθούν κάποια κράτη-μέλη να αντιτίθενται. Αναφέρονται τώρα στο πρόβλημα της επικουρικότητας. Αλλά νομίζω ότι με τη ρήτρα ευελιξίας αυτό έχει ήδη διευθετηθεί. Τώρα, κατά πόσο υπάρχει αρκετή αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών. Όχι, δεν υπάρχει αρκετή αλληλεγγύη, αυτό το γνωρίζουμε και ξέρετε μας αποδυναμώνει αυτό. Διότι οι άνδρες μέσα στις εταιρείε, στα κρατημέλη στην Ευρώπη είναι πολύ καλύτερα διαδικτυωμένοι και δικτυωμένοι. Και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Σε τεφάρ τις μετανάστριες. Το θέμα αυτό της βίας κατά των γυναικών σε κλιματικότητα το έχω θέσει στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης. Και κάλεσα τους Υπουργούς Δικαιοσύνης να προβούν σε όλα τα προληπτικά μέτρα στα κρατη ώστε τα παιδιά και οι γυναίκες να μην πληρώνουν το τίμημα ως ευαίσθητες, ευάλωτες ομάδες. Και βέβαια ε, τα πρώτα θύματα βίας είναι πάντοτε οι πιο αδύναμοι και πιο ευάλωτοι και σίγουρα μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι μετανάστριες. Ε, έτσι λοιπόν πρέπει να δοθεί ε, σημασία και στο προληπτικό σκέλος και όχι μόνο στο σκέλος της καταστολής. Δεν απάντησα τώρα για τη ψηφιακή, τις ψηφιακές τεχνολογίες ICT για τις γυναίκες. Έχω έρθει σε επαφή με ενώσεις που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στον τομέα των και σε ό,τι αφορά ειδικά την ψηφιακή ε, σφαίρα ιδίω για τι ΗΠΑ, ε, βλέπουμε ότι πολλέ θέσει ε, ε, καλύπτονται από γυναίκε. Δηλαδή πολλέ νέες στην αγορά, την ψηφιακή, είναι γυναίκε. Αν έχετε κι εσεί πάντως κάποια ιδέα, ευχαρίστω να την ακούσω. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γιούροβα, σας ευχαριστώ για την ε, ευελιξία που επιδείξατε και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης. Ε, η ώρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι το επόμενο θέμα. Εξαντλήσαμε το χρόνο, άρα θα συζητήσουμε τις εκθέσεις περιαπαλλαγής μετά την ψηφοφορία. Έχετε τις ε, κάρτες για να ψηφίσουμε. Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Τροπολογία 37. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 41, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 51 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική 7 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 57 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 61 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 64 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 65 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές. Α, δεν είμαι βέβαιη. Θα έχουμε λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 16 είναι η ψήφη υπέρ γιατί η κυρία Χάνιμπολ δεν έχει μαζί της την κάρτα της ή κάνω λάθος. Γιατί αλλιώς θα είχαμε ισοψηφία. Άρα εγκρίνεται η κανω λαθος γιατι ελεγε θα ειχαμε ισοψηφια αρα εγκρινεται η τροπολογια το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας. Πάμε στην 66 ψήφη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 67 ψήφι Κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε λοιπόν την τροπολογία 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 68 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71, δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 71 άρχεται η ψηφοφορία. Σε Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 76 ψήφι ΠΕΡ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 77, δύο τμήματα, το πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 77, άρχεται η ψηφοφορία. Θα πρέπει κάποιος ή κάποια από το ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών να βγάλει την κάρτα γιατί είναι υπεράριθμη ομάδα. Ψηφίζουν, ψηφίζει ένας παραπάνω. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Λοιπόν, εγκρίνεται. Πού είμαστε τώρα όμως. Τροπολογία 78. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 79. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 80. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 97 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές να ελέγξουμε τροπολογία υπερθυμών 9 άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας ήταν σαφές. Μάλλον δεν βλέπω καλά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές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 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβεβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ λέω να ελέγξουμε την 33. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Bueno, y Χωρίς όμως άλλη διακοπή, περνάμε στο τελευταίο σημείο της μέρης διάταξης. Ουσιαστικά είναι δύο, αλλά επειδή πρόκειται για την απαλλαγή για το Γενικό Προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν συμφωνείτε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα δύο ε, σημεία μαζί. Η συγκίτρια είναι η ίδια, είναι η κυρία Ματέρα, τη είναι μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις δύο αυτές γνωμοδοτήσεις για την απαλλαγή, γιατί ως Επιτροπή, ως Επιτροπή Γυναικών μας ζητήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να δώσουμε απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το Οικονομικό έτος 2014, αλλά και απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του Γενικού Προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι για το οικονομικό έτος 2014. Ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων προωθεί την ισότητα των φύλων σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απαλλαγή λοιπόν για το 2014 μπορεί να χορηγηθεί, βασισόμαστε εδώ πέρα και σε μια γνωμοδότηση του Ελεκτικού Συνεδρίου, η οποία γνωμοδότηση περιλαμβάνει θετικά στοιχεία όσον αφορά τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Αυτού Ινστιτούτου. Ακόμα και τα μυϊκές ροές για το οικονομικό έτος 2014 δεν παρουσιάζουν παρατυπίες. Παρουσιάζονται μόνο κάποιες καθυστερήσεις όσον αφορά τις πληρωμές και αφαιρούν πιο συγκεκριμένα πιστώσεις επιχειρησιακές και πάλι εδώ πέρα η καθυστέρηση των επιχειρησιακών αυτών πιστώσεων οφείλεται σε συνθήκες εκτός του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Επίσης είναι θετικό ότι υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού λογιστικού ελέγχου για την περίοδο 2015 έω 2017. Δεδομένου λοιπόν ότι δεν υπάρχουν προβληματικά σημεία και ότι γενικά η αποτίμηση των οικονομικών του Ινστιτούτου αυτού ήταν θετική, θεωρούμε ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή για το έτος 2014. Μπορούμε λοιπόν εμείς να στηρίξουμε την ε, έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Προφανώς βέβαια οι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλουν τροπολογίες. 17 Δεκεμβρίου είναι καταληκτική ημερομηνία, 12 το μεσημέρι. Όσον αφορά τώρα τη δεύτερη γνωμοδότηση που έχει να κάνει με την ε, εκτέλεση του Γενικού Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό του 2014 και ιδίω για την πολιτική ισότητα των φύλων της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Ξέρετε ότι εμείς θέλουμε να εντάξουμε τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το 2016 δυστυχώς στο προπολογισμό βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση όσον αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών και την ισότητα των φύλων. Υπό το φως λοιπόν αυτής της μείωσης θα ήθελα να σας πω ότι ε, στο κεφάλαιο του προπολογισμού προβλέπεται για τα δικαιώματα την ε, ηθαγένεια και τη δικαιοσύνη προβλέπονται μειωμένε χρηματοδοτήσεις όσον αφορά το πρόγραμμα Δάφνη, που αποτελεί πλέον στόχο και όχι απλώ πρόγραμμα. Ενθαρρύνουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει πλήρη εφαρμογή του προγράμματος αυτού και πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Δάφνη. Δεν μπορεί να αποδυναμώνεται κατά αυτόν τον τρόπο με περικοπή των πιστώσεων. Λέμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνεται συνεχώς αναφορά στην ενσωμάτωση της διάταξης του φύλου και σε μια κατάρτιση προπολογισμού με γνώμονα την ισότητα των φύλων. Αυτές είναι οι βασικές μας προτεραιότητες Ξέρετε ότι ε, εδώ και πολλά χρόνια είτε ως σκιώδης εισηγήτρια είτε ως εισηγήτρια είχα αναλάβει την ε, απαλλαγή τόσο για τον προπολογισμό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και θεωρώ πλέον ότι έχω δώσει μέσω της γνωμοδότησης αυτής ή των δύο αυτών γνωμοδοτήσεων μια πιο σφαιρική, ολιστική εικόνα των γενικότερων παρατηρήσεων που έχουν εκφράσει κατά καιρού και οι συνάδελφοι στα πλαίσια της α, Επιτροπής αυτής. Και για τη γνωμοδότηση αυτή πάλι καταληκτική ημερομηνία απολογιών είναι 17 Δεκεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Αυτά ήθελα να σας πω. Συγγνώμη αν μίλησα πολύ γρήγορα τους διερμηνείς, αλλά τουλάχιστον τήρησα το χρόνο κόρευση που μου είχατε δώσει, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Ματέρα. Η κυρία Μίλνα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Γρήγορα και σύντομα, επειδή και η συγγήτρια ε, έχει λίγο χρόνο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας και συμφωνώ πλήρως με αυτό που μόλις είπατε. Θα ήθελα και εγώ να αναγνωρίσω ότι η AJ έχει μια αποτελεσματική και σωστή διοίκηση και στην ουσία ε, υποστηρίζει το Ινστιτούτο ε, την δουλειά της Επιτροπής μας. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω την σημασία της συνεργασίας και τα κοινά project που ε, έχουμε. Πρέπει λοιπόν εμείς ε, να είμαστε πλήρως δεσμευμένοι και να χρησιμοποιούμε και τα δεδομένα που δίνονται για μας. Επίσης συμφωνώ με την σημασία τον, ε, του προϋπολογισμού για τα φύλλα. Χρειαζόμαστε τους πόρους ε, ε, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δαπάντες λαμβάνουν υπόψη το φύλλο μέσα από μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την ισότητα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπορσάν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ματέρα για την πολύ σημαντική εργασία της και να την ευχαριστήσω και για αυτό το εξαιρετικό έγγραφο. Να τονίσω ότι το Ινστιτούτο πραγματικά ε, υποστηρίζει πολύ τη δουλειά μας και ε, η εξέταση των οικονομικών του από τα αρμόδιο όργανο δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ε, θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς ε, που, έχουν, δεν έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του Ινστιτούτου. αυτό δεν είναι ε, κάτι που λαμβάνεται θετικά και όσον αφορά όμως την ισότητα των φύλων. Ε, δεν βλέπω να υπάρχουν προβλήματα με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Να πούμε, από μόνοι μας μπορούμε ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά, να δούμε την επίδευξη των στόχων. Και το έχει κωδικοποιήσει αυτό η Κομισιόν Ίνκο και η ΕΝΒΗ επίσης ε, εμπλέκονται και οι πολιτικές που αποφασίζονται εκεί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την ισότητα. Υποστηρίζω πλήρως ε, τη συνάδελφο Μπάρμπαρα και άλλους, αλλά θα ήθελα να υποστηρίξω και τη σημασία των δικτών. Ευχαριστούμε κυρία Φερέντσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο Μπάρμπαρα Ματέρα, η οποία ασχολήθηκε με την εκπόνηση των δύο αυτών γνωμοδοτήσεων εξ ονόματος της δικής μας Επιτροπής θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και ποια είναι η ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Αυτό Ινστιτούτο. Χαίρομαι πάρα πολύ που στο σημείο 7 της γνωμοδότης αναφέρεστε στην ενίσχυση και περαιτέρω συνέχιση αυτής της συνεργασίας. Λέτε επίση ότι εκτελέστηκε σωστά ο προπολογισμό από το Ινστιτούτο αυτό. Θεωρώ ότι την άποψη αυτή θα έχει και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Θα ήθελα να πω επίσης ότι το Ινστιτούτο αυτό έχει δεσμευτεί όχι μόνο να συνεργάζεται με τη δική μα Επιτροπή, αλλά εν γέννη να συνεργάζεται για το ζήτημα του gender mainstreaming με όλες τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι η συνεργασία αυτή για την ενσωμάτωση διάσταση του φύλου είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, ξέρετε ότι τα Ηνωμένα Έθνη μας ζητούν να καταφέρουμε να πετύχουμε μέχρι το 2030 μια απόλυτη ισότητα των δύο φύλων. Να κάνω όμως και μια παρατήρηση. Όχι μόνο συμφωνώ προφανώς με τα όσα έχουν να κάνουν με το λεγόμενο gender budgeting, ε, εκπόνηση προπολογισμού με γνώμονα την ισότητα των φύλων, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερο οι δείκτες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων. Άλλωστε αυτό το συστήσαμε πριν από λίγο και με την Επίτροπο. Εγώ ήρθα σε επαφή με την ε, πρόεδρο του Ιταλικού Κοινοβουλίου και είπα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ του Ιταλικού Κοινοβουλίου καθώς επίσης και της Εθνικής Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας προκειμένου να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα για τις γυναίκες σε περιφερειακό επίπεδο. Κυρία Μορβά, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για θέματα ισότητας ε, πόσο ψηλό προπολογισμό έχει. Ε, είμαι έξι χρόνια βουλευτής και στο μεταξύ έγινα και μέλος αυτής της επιτροπής. Παίρνουμε έτσι ένα τετράδιο στα χέρια, αλλά στην ουσία τι output έχουμε. Ε, με αυτό το ψηλό προϋπολογισμό, ε, τι βγάζει αυτό το Ινστιτούτο γενικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις ε, Ευρωπαίες γυναίκες. Μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο γι' αυτό. Το ερώτημα είναι το ίδιο και για το πρόγραμμα Δάφνη. Έχει γίνει στην ουσία ένας κλάδος ε, που προσπαθεί να πατάξει τη βία. Όμως ε, δεν στοχεύει τα θύματα, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που συνεχώς ε, ασκούν αυτή τη βία. Υπάρχει μια ιδεολογία πίσω από αυτό και δεν δίνεται καμία βοήθεια στα θύματα, στις γυναίκες. Ε, υπάρχει κακοποίηση των γυναικών, ξυλοδαρμός και τόσα χρήματα δίνονται για αυτό. Ποια είναι τα αποτελέσματα. Και για να κλείσουμε αυτό τον ε, γύρο η κυρία Βάνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ματέρα για την εξαιρετική γνωμοδότησή της εκ μέρους της δικής μας ομάδας. Η γνωμοδότηση για την ΑΕΚΙΕ δεν έχει κάτι παραπάνω ε, για μένα που πρέπει να σχολιαστεί, πέρα από αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι και εγώ θεωρώ ότι το ΕΓΕ μας υποστηρίζει στη δουλειά μας και θα ήθελα ε, κι άλλο προσωπικό που θα ήταν απαραίτητο Τώρα όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2016 θα 14, συγγνώμη, ε, θα πρέπει το gender budgeting που έχει ήδη υποθεί από τους συναδέλφους ε, να ληφθεί υπόψη και στο αποτελεκτικό ε, συμβούλιο, να λάβει δηλαδή υπόψη του το συμβούλιο πόσο σημαντικό είναι το θέμα της ισότητας των φύλων. Σας ευχαριστούμε κυρία Βάνα και για να κλείσουμε αυτό το σημείο της μερσιάς διάταξης μετά τις παρεμβάσεις των συναδέλφων θα δώσω για μια ακόμη φορά το λόγο στην κυρία Ματέρα. Αγαπητοί συνάδελφοί, σας ευχαριστώ πολύ γιατί συνήθως πλήττει κανείς όταν συζητάμε ζητήματα προπολογισμού, ενώ εσείς θίξετε ζητήματα τα οποία είναι άκρος ενδιαφέροντα. Άκουσα λοιπόν αυτά που είπε η κυρία Βάνα και θα τα λάβω όλα υπόψη μου. Νομίζω ότι θα πρέπει κυρίως να διαβάσετε και τα κείμενα αυτά, τα πάντα αναφέρονται προβλέπονται 7 εκατομμύρια ευρώ για το ΑΕΓΕ. Είναι πολύ σημαντικό το Ινστιτούτο αυτό. Πρέπει να σας πω όμως ότι ε, μολονότι είμαι αρκετά νέα, είμαι 7 χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να σας πω ότι από τότε που ιδρύθηκε το Ινστιτούτο αυτό, πριν από μερικά χρόνια, πραγματικά η συμβολή του είναι πάρα πολύ σημαντική ουσιαστικά προωθεί πολιτικέ ισότητα των φύλων παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλε τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στάση του λοιπόν θεωρώ ότι είναι επικοδομητική. Νομίζω λοιπόν ότι αν διαβάσετε λίγο τα σχετικά έγγραφα θα βρείτε απαντήσει για τη χρησιμότητα του Ινστιτούτου αυτού. Σας ευχαριστώ κυρία Ματέρα. Όπως ε, είπε λοιπόν ε, η κυρία Ματέρα, έχουμε ως προθεσμία τη 17η Δεκεμβρίου για την κατάθεση τροπολογιών. Όταν λοιπόν ε, μάλλον λίγη εδώ η συνεδρία, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και σας εύχομαι ένα καλό βράδυ.